Έχουν κατατεθεί έξι ψηφίσματα συνολικά για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, η οποία και ολοκληρώνεται και περνούμε μέσω στι ψηφοφορίε. Αρχίζουμε με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πέντε πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει ψήφισμα. Ε, τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά, επίσης απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο ψήφισμα που αφορά την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα. Πέντε πολιτικές ομάδες. Τμήμα πρώτο της παραγράφου 3 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές επίσης εγκρίνεται. Παράγραφος 6, τροπολογία 2, ψήφι πέρα. Κατά. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται τελογική σκέψη F, ε, τοπολογία 1 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφιζόντος όπως πείθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τελευταίο ψήφισμα κατάσταση στη Σρι Λάνκα. Και εδώ έχουμε λάβει ένα ψήφισμα κοινό πέντε πολιτικών ομάδων. Μετά την παράγραφο 1, η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, επίσης απορρίπτεται. Παράγραφος 9 το αρχηγού κειμένου σε δύο τμήματα και τα δύο νομιμαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα και πάλι ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι μου. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 ψήφι υπέρ. Κατά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Την ε, τροπολογία 3 αρχίζει τώρα. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 4 ψηφίπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τα πρακτικά, τα συνοπτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση την επόμενη φορά και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ε, τα ψηφίσματα που μόλις εγκρίναμε θα τα διαβιβάσουμε στους ε, αποδέκτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνει εδώ μια ε, μακρά χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ.